και τη Νέα Ζηλανδία. Το λόγο έχει για πέντε λεπτά ο κύριος Λάγκε, συντάκτης της ερώτησης. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι συναδελφοί, κύριε Επίτροπε. Ακούσαμε και διαβάσαμε σχετικά με την εμπορική στρατηγική ότι θα έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και ο χώρος της, ε, ε, του ειρηνικού στην, ε, στις εμπορικές μας σχέσεις. Και εν ώψη της συμφωνίας του ειρηνικού πολιτειών με 11 εταίρους τους, βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία παίρνει. Πρόκειται για το τρίπλο π. Είναι λογικό λοιπόν δεδομένων και των σχέσεων που έχουμε με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία να στραφούμε και εμείς προς την ίδια κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έκανε μία συνάντηση τύπου workshop για να μελετήσει το ζήτημα αυτό και έτσι προχωρούμε με τη συμφωνία ε, με τη συζήτηση καλύτερα της συμφωνίας για ε, εμπορικές σχέσεις με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Βεβαίω έχουμε πολύ στενές σχέσεις με τις χώρες αυτές, κοινότητα αξιών πάνω απ' όλα, δημοκρατικές δομές και αντίστοιχες οικονομικές τοποθετήσεις. Άρα έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Η Αυστραλία είναι στην 21η θέση κρατών όπως η Νέα Ζηλανδία στην 51η κρατών σε όγκο εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι χωρισμένα είναι σε πρώτες θέσεις, είναι πάντως σε όχι ασήμαντη θέση και σημασία. Από την άλλη έχουν πολύ σημαντικούς τομείς, γεωργικό, γάλα και ζάχαρη, όπου έχει γίνει πολύ εντατική συζήτηση, ε, παραγωγή, παραγωγή κρέατος και τα θέματα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ε, πρόβιο κρέας ιδιαίτερος, προέλευση γεωγραφική και ονομασία προελεύσεως που αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τη μία και την άλλη πλευρά, την Ευρώπη δηλαδή και την Αυστραλία. Υπάρχουν διαφορές λοιπόν. Αλλά προχωρούμε προς την εγκαθίδρυση κοινών κανόνων. Και αυτό είναι λογικό δεδομένης και της προόδου της υφηλίου προς την παγκοσμιοποίηση οι κανόνες αυτοί είναι καλύτερο βεβαίως να αναπτυχθούν με χώρες οι οποίες έχουν αντίστοιχες θεωρήσεις, αντίστοιχες δημοκρατικές δομές και γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι όταν συνομιλούμε με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία μπορούμε να μιλάμε με πολύ, να διατυπώνουμε πολύ πιο φιλόδοξες απαιτήσει από ό,τι έκαναν οι Αμερικανοί στην αντίστοιχη συμφωνία πέραν του ειρηνικού. Μπορούμε επίσης να κάνουμε ανάλυση των ε, κερδών και των συνεπειών τέτοιων συμφωνιών. Και κυρίως θα ήθελα να επιμείνω στο θέμα του δυναμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε, περιμένω να μας εκθέσετε τις απόψεις σας, γιατί πρώτη φορά συνέβη φέτος να περιοριστεί, να συρρυκνωθεί ο αριθμός του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Trade για το Διεθνές Εμπόριο. Δεν νομίζω ότι είναι η εποχή τώρα να περικόπτουμε σε αυτούς τους τομείς την υποστήριξη που προσφέρουμε. Χρειάζεται, γιατί είναι πολύ σημαντική, όλο και σημαντικότερη η πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να υπάρχει επαρκής επάνδρωση. Ταυτόχρονα χρειάζεται διαφάνεια, ταυτόχρονα χρειάζεται σαφήνεια, γι' αυτό έχουμε διατυπώσει και προφορική ερώτηση που περιμένουμε ε, να συμπληρώσουμε με την δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου, ερώτηση που διατυπώνει το γιατί τώρα αυτή η συμφωνία ή τι είδους κίνδυνοι μπορεί να προκύπτουν από αυτή τη συμφωνία, τι συνέπειες μπορεί να έχει και για το χώρο του ειρηνικού, η συμφωνία με την Αυστραλία και, τη Ζηλανδία, όπου και την Αζηλανδία, όπως επίσης τι χρονικό ε, διάγραμμα βλέπετε στη συμφωνία αυτή. Αυτά θα περιμένουμε ως απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Λάγκε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μίμητσα. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία είναι δύο εταίροι που είναι σαν την Ευρώπη, με τους οποίους έχουμε τόσες κοινέ αξίες. Η ενίσχυση των σχέσεων μαζί τους λοιπόν αποτελεί προτεραιότητα για μας. Και γι' αυτό το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε διαπραγματεύσεις για ε, πολιτικού πλαισίου συμφωνίες τόσο με την Αυστραλία όσο και με την Νέα Ζηλανδία προκειμένου να ενισχύσουμε καλύτερα την εταιρική μας σχέση μαζί τους επειδή ακριβώ έχουμε κοινέ αξίες όπως είναι σεβασμός δημοκρατικών αρχών, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες, κράτος δικαίου και η προώθηση της ειρήνης στον κόσμο και της ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λοιπόν σχέσεις όριμες όσον αφορά το εμπόριο με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής, ο μεγαλύτερος εταίρος όσον αφορά τις υπηρεσίες της Αυστραλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών για τη Νέα Ζηλανδία, αλλά και υπηρεσιών και δεύτερος όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, λοιπόν, έχουν με την Κίνα, το ΑΣΕΑΝ, την Ιαπωνία, την Κορία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και πρόσφατα και με τον Ειρηνικό. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς εμπορικών αγαθών, ε, υπηρεσιών κτλ. βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση από ό,τι οι ανταγωνιστές τους. Στην πράξη, τα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι τα μόνα που θα πληρώνουν τέλη στην Αυστραλία για την εισαγωγή τους εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Αυστραλία και ο δεύτερος στην Νέα Ζηλανδία. Όμως οι Κινέζοι επενδυτές έχουν πιο εύκολη πρόσβαση τόσο στην Αυστραλία όσο και στη Νέα Ζηλανδία εξαιτία αυτών των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και συμφέροντα επίσης στον τομέα των κρατικών προμηθειών. Και θέλουμε να ενισχυθούν τα δικαιώματα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας στον ΠΟΕ. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, γαλακτοκομικά, βόλιο κρέας, πρόβιο κρέας και ζάχαρη. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλες ευαισθησίες στον τομέα αυτό, όπως είναι η Ιαπωνία και η Κορέα, κατάφεραν να έχουν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, λέγοντας ότι τέτοια ευαίσθητα ζητήματα μπορούν να τα διαχειριστούν τελικά. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εποφελούνται και οι δύο από προτιμησιακή πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα ευαίσθητα προϊόντα επειδή υπάρχουν ποσοστώσεις. Όσον αφορά τώρα τις γεωγραφικές ενδείξεις, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετική από εκείνη της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι θα θέσει ενισχύ για το κρασί και τα ενοπνευματόδη τη γεωγραφική ένδειξη για την Αυστραλία έχουμε ήδη μια συμφωνία για τον Ίνο με γεωγραφικές ενδείξεις. Θέλουμε πλήρη προστασία της γεωγραφικής ένδειξης, όχι μόνο στον Ίνο και τα ενοπνευματόδη, αλλά και στα τρόφιμα γενικά. Οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου δίνουν την ευκαιρία να εξευρεθούν λύσεις. Συνεπώς. Σε πρόσφατες συναντήσεις ανάμεσα στην Προεδρία της Επιτροπής και του Συμβουλίου με τον Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας τον Οκτώβριο που μας πέρασε και με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας τον Νοέμβριο, υπήρξε συμφωνία για να αρχίσουν οι εργασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις δύο αυτές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τη μελέτη της αντικτύπου με διαβούλευση με το κοινό και διμερώς θα γίνουν μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα αυτά θα ολοκληρωθούν πριν ζητήσει η Επιτροπή την άδεια από το Συμβούλιο για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρατά ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ΙΝΤΑ, την Επιτροπή και την Ομάδα Εργασίας για τη Νέα Ζηλανδία όσον αφορά τις εξελίξεις προχωρώντας αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ξέρετε ότι έχουμε μια κάποια καθυστέρηση. Θα πρέπει να σεβαστείτε το χρόνο ομιλία σας. Ο κύριος Κάσπαρη έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε το θέμα της Αυστραλίας και της Ελληνικής και της σχετικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Είναι λίγα τα μέλη του ΠΟΕ με τα οποία δεν διαπραγματευόμαστε ή δεν έχουμε συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Από αυτά η Αυστραλία και η Νέα κράτη με τα οποία έχουμε κοινέ αξίες και δομέ είναι κράτη με τα οποία πρέπει να να αναπτύξουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και ταυτόχρονα πολλά κράτη της περιοχής έχουν μαζί μας ή έχουμε εμείς με τα κράτη αυτά ε, συμφωνίες. Έχουμε ήδη συνάψει με την Νότια Κορέα, είμαστε σε διαπραγμάτευση με την Ιαπωνία και αντίστοιχες άλλες χώρες. Μιλούμε για επενδυτικές συμφωνίες με την ε, Κίνα. Είναι κατεπίγουσα λοιπόν η ανάγκη για μένα να προχωρήσουμε σε μια γερή βάση, ε, συμβατική βάση για τις εμπορικές συναλλαγές με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Θα ήθελα πριν από την ανάθεση βέβαια των εντολών να είμαστε βέβαιοι, της εντολής, να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Είναι πολύ σωστό να ξεκινούμε το ταχύτερο δυνατό ε, ως προς την επισήμανση των δικών μας οικονομικών συμφερόντων, την επιθετική αυτή δηλαδή επιχειρηματική. Ε, διαπραγματευτική στρατηγική, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και προβλήματα, επιθυμίες αλλά και ανησυχίες που εκδηλώθηκαν πρόσφατα ιδιαίτερα στην ε, Γεω, στον τομέα της γεωργίας, τις πιο απομακρυσμένες κυρίως περιοχές της Ευρώπης και θα πρέπει και αυτά να τα επισημάνουμε και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την ε, υποχωρήγηση εντολή που ζητάτε τι έχετε να απαντήσετε σε σχέση με τις ανησυχίες και τα μελήματα που έχουν εκφραστεί και βέβαια εμείς από το Κοινοβούλιο θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή την εντολή που βέβαια θα πρέπει να εγκριθεί και από το Συμβούλιο. Εκ μέρους των Σελιστών και Δημοκρατών, Κράς Βάντερ Χάιντς. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Αυτή η συμφωνία με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία δεν μπορεί να αποτελέσει αυτό σκοπό. Επουδενή πρέπει να αποτελέσει μέσον για την υλοποίηση ενό στόχου. Πρέπει δηλαδή να προσφέρει πλεονεκτήματα για τον πολίτη, άντρα και γυναίκα. Χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη να φέρει, χρειάζεται δηλαδή να βελτιώσει τι ευκαιρίε για δημιουργία θέσεων εργασία. Και πάνω απ' όλα δεν μπορούν να υποβαθμιστούν ε, οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστασία της υγείας ή για τις δημόσιες υπηρεσίες, την πνευματική ιδιοκτησία, τη γεωγραφική προέλευση και πάνω απ' όλα ο τομέας της γεωργίας που είναι από τους πιο ευάλωτους θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προστασίας. Η διαφύλαξη των κοινωνικών και εργατικών προδιαγραφών έχει ύψιστη προτεραιότητα για μας. Εδώ δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τον παραμικρό συμβασμό και γι' αυτό απαιτούμε ένα ε, φιλόδοξο κεφάλαιο για την αηφορία. Όπως και, σε άλλες πολλές, όπως και άλλοι πολλοί συνάδελφοι θέλουμε διαφανείς διαπραγματεύσεις και συμμετοχή και τη κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ. Μακλάρκιν, ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έχει την ευκαιρία τώρα για τα επόμενα χρόνια να διαπραγματευτεί μια σύγχρονη συμφωνία εμπορικών συναλλαγών για τον 21ο αιώνα με εταίρους που ομονοούν την ε, Αυστραλία και την Ζηλανδία, που ομονοούν μαζί μας, που έχουμε αντίστοιχες αξίες, που έχουμε ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, χώρες που είναι στρατευμένες και προσυλλομένες και στην πολυμερή, στο πολυμερές θεματολόγιο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και βέβαια ταυτόχρονα θέλουν να ανοίξουν εμπορικές αγορές σε διμέρες επίπεδο ώστε να δώσουν και άλλες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των σχέσεων τους με την περιοχή της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού. Έχουμε θέματα για τις γεωργικές, για τις ονομασίες ε, προελεύσεως, για την προστασία των προϊόντων μας. Έχουμε πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης εμπορικής ε, συμφωνίας που θα λύσει προβλήματα της σύγχρονης εποχής, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ψηφιακή οικονομία και βέβαια θα προβλέπει και κεφάλαιο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επωφελούνται τα μάλα από τις εμπορικές συμφωνίες. Εγώ θα υποστηρίξω τις επραγματεύσεις αυτές και πιστεύω ότι μπορούμε το χέτερο δυνατόν να τις ολοκληρώσουμε. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Ο κύριος Τάκουλα, δύο λεπτά. Φιλελεύθερη. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την προφορική ερώτηση για την Επιτροπή και το ψήφισμα της Επιτροπής ΙΝΤΑ και τα εξετάζουμε μαζί σήμερα στα πλαίσια της έναρξης διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται τέτοιε συμφωνίε με πολλέ τρίτε χώρε και δημιουργεί έτσι σταθερέ οικονομικέ σχέσει και οικονομική ανάπτυξη για μα και του άλλου κάτι που μας θωρακίζει σε περίπτωση αστάθειας. Αλλά έχουμε μείνει πολύ πίσω, δεδομένου ότι δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τέτοιες συμφωνίες με μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίες οικονομίες στην Αυστραλία. Και αυτό μας εκπλήσει, γιατί παραδοσιακά έχουμε σχέσεις και με την Αυστραλία και με τη Νέα Ζηλανδία σε πολλούς τομείς και πιστεύουμε στις ίδιες κοινέ αξίες. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να μείνουμε εκτός του κύκλου αυτού που χτίζεται γύρω από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Ενδυναμώνοντας λοιπόν τη συνεργασία μας και πηγαίνοντας περισσότερο σε βάθος τις σχέσεις μας με αυτές τις χώρες, μπορούμε έτσι να προωθήσουμε δίκαιες αρχές προστατεύοντας τους σπόρους. Γι' αυτό λοιπόν ρωτάω, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρχίσει ακόμα διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Αυστρία και η Νέα Ζηλανδία έχουν δηλώσει ότι θέλουν να αρχίσει αυτή η διαδικασία και είμαι πεπισμένο ότι όλες αυτές οι χώρες θα υποφεληθούν από μια τέτοια συμφωνία όπως έχει συμβεί και με όλες τις άλλες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που έχουμε διαπραγματευτεί μέχρι τώρα. Συνεπώς, κάνω έκκληση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει το σκόπιγο όσο γίνεται πιο γρήγορα και να δεσμευτεί ότι θα περάσει στο επόμενο βήμα διαπραγματεύσεων για αυτήν την αμοιβαία υποφελή ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Για ένα λεπτό τώρα εκ μέρου της Γκουέ Σάντσες Καλντεντέι. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργείται ένα είδος ε, δόγματος πάνω στο οποίο ε, τυφλά εμένουμε χωρίς ε, να λαμβάνουμε υπόψη μας τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σε επίπεδο εσωτερικής ζήτησης. Το ίδιο συμβαίνει και με τις συμφωνίες αυτές τις εμπορικές και με τις, τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία την ειδική στην περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας ε, θα πρέπει να υπογράψουμε μια συμφωνία αλλά να έχει προοπτική, να μην εμένει σε δογματικές αντιλήψεις, να δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους, σε ποιο βαθμό μπορεί να ενισχύσει το σεβασμό του περιβάλλοντος και την προστασία του περιβάλλοντος ανάμεσα στις τρεις συμβαλόμενες πλευρές. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και να υπερασπιστούμε ε, τα δικαιώματα του ίδιου του πλανήτη. Κυρία Χόιμπουχ, μισή λεπτό, πράσινη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Τα, γεωργα... τα αγροτικά προϊόντα είναι πολύ σημαντικά δεξαγωγικά προϊόντα και για την Αυστραλία και για την Νέα Ζηλανδία και γι' αυτό το δυναμικό μια συμφωνία εμπορικών συναλλαγών με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία θα πρέπει ιδιαίτερα να θέσει τη γεωργία στο επικέντρο των συζητήσεων. Αλλά δυστυχώ στην πρόταση ψηφίσματο αυτό δεν επισημαίνεται. Επαρκώ η παραγωγή και το κόστο παραγωγή γάλακτο στην ε, Νέα Ζηλανδία. είναι πολύ σημαντικότερη, πολύ χαμηλότερη από ότι εδώ. Σε εμά στη Γερμανία, παραδείγματι, είναι 10 λεπτά του ευρώ, ακριβότερο το λίτρο του γάλακτος. Το ίδιο συμβαίνει και με το, βόιο, με το πρόβιο κρέας, τη ζάχαρη και άλλα προϊόντα. Οι γεωργοί μας διαμαρτύρονται, δεν εισπράττουν αρκετά χρήματα και λόγω της ε, ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό δεν έχουν επαρκή έσοδα και θεωρούν ότι τα προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να διαθέσουν στην αγορά ε, είναι πολύ φθηνότερο να μην τα παράγουν καν. Οι Ευρωπαίοι Γεωργοί λοιπόν θα, έρθουν σε άμε... θα βρεθούν αντιμέτωποι απευθείας με τον ανταγωνισμό των Αυστραλών και Νεοζηλανδών Γεωργών. Είναι σαν να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά λοιπόν. Πρέπει να βγει το γάλα από το τομέα των διαπραγματεύσεων και πρέπει οι αρνητικές συνέπειες από την ε, ανταλλαγή γεωργικών προϊόντων να ε, αντιμετωπιστούν. Δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε προϊόντα σε όλο κλήρο τον κόσμο, προϊόντα τα οποία ούτως ή άλλως παράγουμε εδώ και πρέπει να μείνουν εδώ. Ευχαριστώ Μπέγκιν. Ένα λεπτό η παραγουμε εδω και πρεπει Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το να ε, ανοίγουμε διαπραγματεύσεις με χώρες ε, μακρινές όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχει να κάνει με την προσπάθεια να ε, αναπτύξουμε εμπορικές συναλλαγές σε αγορές που θα συμπληρώσουν αυτή τη συμφωνία της ε, διατλαντικής ε, σχέσης και θα ήθελα να αναφερθώ στις απειλές που επεσήμαναν και άλλοι συνάδελφοι, απειλές ε, που μπορεί να επηρεάσουν και οι γεωπολιτικές μας επιλογές. Δεν μπορούμε να έχουμε μία συμφωνία αν δεν λάβουμε υπόψη και τις διαιτερότητες και τα προβλήματα του γαλακτοκομικού τομέα. Έχουμε ήδη πολλά προβλήματα εκεί. Έχουμε ήδη πολλά προβλήματα ως προς τις ε, ονομασίες προελεύσεως ε, με τη συμφωνία αυτή. Χρειάζεται διαφάνεια λοιπόν, χρειάζεται σαφήνεια και πάνω απ' όλα διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις. Ήδη μας έχει αποδειχθεί ότι, και από προηγούμενες συμφωνίες ότι πρέπει να σεβόμαστε τους πολίτες και τις επιλογές τους. Η φωνή των πολιτών λοιπόν θα ακουστεί και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Φέλνερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η συμφωνία αυτή ελεύθερων συναλλαγών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι δύο από τις έξι χώρες με τις οποίες δεν έχουμε ακόμα τέτοιου είδους συμφωνίες. Οι άλλες είναι η Βόρεια Κορέα, η Κορέα, η Ρωσία και η Ταϊουάν. Η Αυστραλία λοιπόν και η Νέα Ζηλανδία βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε μας όμως. Οι συμφωνίες, συνεπώς, ελεύθερων συναλλαγών θα βοηθήσουν να μην βγει χαμένη η Ευρώπη. Υπάρχουν βέβαια προϋποθέσεις που πρέπει να υποστηρίξουμε. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδειχτεί φιλόδοξη όσον αφορά τους κανόνες που τελικά θα διαπραγματευτούμε. Πρέπει να αρχίσουμε ήδη με παγκόσμιες προδιαγραφές. Η Ευρώπη όμως θα πρέπει να ηγηθεί σε αυτή την προσπάθεια. Ήδη υπάρχουν ε, δυσκολίες. Για παράδειγμα όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εξάγουν γεωργικά προϊόντα. Εμείς βρισκόμαστε στην άλλη άκρη του πλανήτη. Κινδυνεύουμε λοιπόν να χάσουμε από τέτοιες συμφωνίες αν δεν προσέξουμε. Δύο πράγματα λοιπόν ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, η συμφωνία αυτή πρέπει να επιτρέψει να εκπονηθούν νέες προδιαγραφές. Και το άλλο που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν πρέπει να σταματήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μαρτίν, ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και εγώ καλώς ορίζω θερμά τι Προθέσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Άνοξη διαπραγματεύσεων για αυτές τις δύο συμφωνίες ελεύθερου εμπολίου. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία αντιστοιχούν σε πολύ ψηλά ποσοστά εμπορικού όγκου για μας. Έχουμε ιστορικούς δεσμούς, είναι πολύ κοντά στον υπόλοιπο χώρο της ασιατικής αγοράς, μπορεί να αποτελέσουν λοιπόν πολύ σημαντικούς εταίρους για μας δεδομένων των εμπειριών από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, αυτές οι συμφωνίες μπορούν να, έχουν, να λάβουν υποδειγματικό χαρακτήρα, μπορούν να προχωρήσουν ταχύτατα και αποτελεσματικά, κάτι το οποίο, δεν έχουμε δει σε σχέση με άλλες εμπορικές συναλλαγές. Μπορούν να αναπτύξουν ύψιστη ποιότητα με κεφάλαιο αηφορίας και ε, παραπομπές σε σχέση με τη λυπή Νοτιοανατολική Ασία και το χώρο του ειρηνικού. Πρέπει ιδιαίτερα να κοιτάξουμε τις ε, την αντιμετώπιση των ροών σε διαφωνίες ή διαφορές για τη που πρέπει να διαφερθούν μεταξύ επενδυτών και κρατών και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν μέσα στις συμφωνίες. Κύριε Μαρτίνα, δέχεστε μία μπλε κάρτα από την κυρία Κάρτενμπαχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Μάρτιν, κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση είχε εκφράσει τις επιθυμίες να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη σχετική έρευνα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιστεύετε λοιπόν ότι αν βγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί αυτό να βλάψει τις σχέσεις μας εμπορικές με τους παλαιούς φίλους και συμμάχους Αυστραλία και Νέα Ισλανδία. Μάρτιν. Βεβαίως. Κάποιοι μάλιστα εδώ λένε ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια εναλλακτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με τα χώρες που ανήκαν στο παρελθόν στην Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία. Αυτό Ωστόσο, νομίζω ότι δεν θα είναι η καλύτερη λύση. Πρέπει να κοιτάξουμε ότι οι χώρε αυτέ έχουν προ το συμφέρον να έχουν συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω αυτή και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και σε αυτό θα πρέπει να, ενθαρρύνουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο Ζαχράντη, λέει ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολείπεται σε ό,τι αφορά την σύναψη συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με τη ζώνη της από Ανατολής και του Ειρηνικού. Άλλες χώρες βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από εμά. Υπάρχουν συμφωνίες που ξεπερνούν τις δικές μας. Εμείς έχουμε απλώ συμφωνίες με την Ιαπωνία η οποία ακόμα δεν έχει κυρωθεί και περιμένουμε ακόμα να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Έχουμε μια συμφωνία με τη Σιγκαπούρη η οποία είναι παγωμένη και περιμένουμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τίποτα δεν έχουμε σε τελική ανάλυση. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον μας να διευρύνουμε τη δυνατότητα του να έχουμε νέες συμφωνίες που θα ανοίξουν αγορές σε μας, όπως της Αυστραλίας και της Νέας Ιλανδίας. Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν λοιπόν. Πρέπει να σπάσουμε τον κύκλο της ιοπής, γι' αυτό εγώ χαιρετίζω αυτές τις προσπάθειες και ελπίζω ότι θα μας φέρουν σε μια ταχεία συμφωνία. Ο Μαρτζή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με την κυρία Μάλστρομ για τα θέματα της προστασίας των ευαισθητών προϊόντων από υπερφερειακές χώρες και περιοχές στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών. <clears throat> Και υπενθυμίζω την δέσμευση που ανέλαβε η κυρία Επίτροπος να φροντίσει το θέμα αυτό ενώπιον των ε, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε λοιπόν πρώτων πυλών της ε, έναρξης διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και ζητούμε από την Κομισιόν και πάλι να κάνει τα απαραίτητα για να προστατευτούν τα ειδικά σάχαρα από τις υπερπεριφερειακές περιοχές που θα μπορούσαν να φυγούν από τις συμφωνίες αυτές και ζητούμε από την Κομισιόν να τηρήσει τα υπεσχημένα. Μόργανο για ένα λεπτό. η Αυστραλία και η Νέα Ισλανδία είναι μόνο γεωγραφικά μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί συμμεριζόμαστε τις ίδιες δημοκρατικές ε, αξίες και αξίες και αρχές που μας συνδέουν. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε αυτή την στενή συνεργασία και σε εμπορικό επίπεδο. Το Φεβρουάριο η αντιπροσωπεία Αυστραλίας Αυστραλίας-Νέα Ισλανδίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω μετέβη στην Αυστραλία. Συναντήσαμε υψηλού αξιωματούχου, αλλά και εκπροσώπους του οικονομικού χώρου. Επομένω, όταν μαθαίνω ότι η Κομισιόν έχει την πρόθεση να ξεκινήσει συζητήσει για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τι δύο χώρε. χαίρομαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σύγχρονε αλλά και εξισορροπημένε συμφωνίε που λαμβάνουν υπόψη τη σημασία ορισμένων τομέων της γεωργικής παραγωγής που έχουν ε, ονομασία προέλευσης και με τον τρόπο αυτό να διευρύνουμε και να ενισχύσουμε το γεωπολιτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λεκάνη του ειρηνικού αλλά να δώσουμε και περισσότερες ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές εταιρείες και με θετικά αποτελέσματα και για τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης. Κυρία Εφώστερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ως αντιπρόεδρο της, ε, της για την Αυστραλία Νέα Ισλανδία. Χαίρομαι για τη σημερινή συζήτηση και χαίρομαι για τα θετικά νέα ότι έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με στόχο να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία με την Αυστραλία αλλά και την Νέα Ισλανδία. Οι συζητήσει αυτέ έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από πολύ παλιά για λόγους προστατευτισμού, για λόγους άσχετους έχουν εμποδιστεί από ορισμένα κρατημέλη και από ορισμένου κοινοβουλευτικούς στην αίθουσα αυτή για να εμποδίσουν την πρόοδο. Σε κάποιο επίπεδο υπήρξε ακόμα και ε, διαφυσβήτηση του ιστορικού των χωρών αυτών στα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο είναι ένα έσχος. Χιλιάδες στρατιώτες από τις χώρες αυτές πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους τον 20ο αιώνα για να απελευθερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Περιμένω κύριε ε, Επίτροπε, ότι θα συνεχίσουν αυτές οι ε, συνομιλίες και θα μπορέσουν να καρποφορήσουν πολύ σύντομα. Αυτό είναι μια κατάσταση win-win για όλους και ελπίζω ότι θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Μορέλ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ακούω τους συναδέλφους που μας λένε τόσα για τις Ηνωμένε Πολιτείες που πρόσφατα, πρόσφατα ε, έκαναν πιο ήπια τη θέση τους για την κατάσταση στον ελληνικό. Εγώ θα έλεγα να είμαστε πάντοτε συνετοί, διότι μπορεί να έχουμε κοινέ αξίες με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία, κυρίως για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την δημοκρατία, όμως έχουμε και πραγματικές διαφορές ως προς την εμπορική μας νοοτροπία. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία αγνοούν την ε, έννοια της γεωγραφικής ένδειξη ω προ τι υπηρεσίε. δεν ε, αποφεύγουν τις ε, αρνητικές, τους αρνητικούς καταλόγους, τις αρνητικές λίστες, ενώ εμείς προτιμούμε τους θετικούς. Όταν λένε λοιπόν οι συνάδελφοι εδώ ότι έχουμε μια συμφωνία win-win με κέρδη για όλους, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ε, να κοιτάξουμε αυτό το άνοιγμα προς την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία και να είμαστε λίγο πιο συνετοί. Είναι λιγότερο περιοριστικοί κανόνες της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας είναι πολύ βιομηχανοποιημένε και εντατικέ εμπορικά χώρε. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τι θα γίνει στην Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Μορέλ, έχουμε πέντε λεπτά για την διαδικασία Κατστιά. Η κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και σας, ε, Επίτροπε, για τις αναρτήρες παρατηρήσεις σας. Πολλοί ανέφεραν το γεωργικό τομέα ως ιδιαίτερα ευαίσθητο και θα ήθελα να μου πείτε περισσότερε λεπτομέρειε για το πώ θα το χειριστείτε αυτό στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι όλα θα, όλες αυτές οι συμφωνίες θα έχουν ωφέλη για όλους, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και όλες οι ιδιαίτερες ευαισθησίες. Υπάρχει και μια μεγαλύτερη όμως ε, ερώτηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιες εμπορικές διαπραγματεύσεις έχει ολοκληρώσει την πορεία, σε κάποιες άλλες ε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ποιο παρακολουθεί το συνολικό πλαίσιο αυτών των συμφωνιών που είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων ταυτόχρονα. Ε, εφόσον ο αντίκτυπο στον γεωργικό τομέα μπορεί να είναι σημαντικό. Το είναι και οι συνάδελφοι. Έχουμε κοινή αγροτική πολιτική, έχουμε πολύ διαφορετική διάρθρωση τη γεωργία στην Ευρώπη. Θέλουμε να παραμείνει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ζωντανή. Πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό και πώ θα γίνει αυτό την πληθώρα εμπορικών συμφωνιών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση στον γεωργικό τομέα συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε κύριο Καπούτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχουν κοινέ αξίε δημοκρατικέ και έχουν την ίδια άποψη για παγκόσμια θέματα ιδιαίτερα επίκαιρα, όπω τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία του περιβάλλοντο, η ανάπτυξη. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί είναι λίγα από τα ε, μέλη του ΠΟΕ. Κύριε Καπούτο, διακόπτη πρόεδρο. λίγο πιο σιγά σας παρακαλούμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν έχει προτιμησιακή πρόσβαση σε, κάποιες, ε, σε κάποια μερίδια της αγοράς των χωρών αυτών. Αυτό δεν έχει νόημα. Σε χώρες όπως Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία υπάρχουν τομείς που είναι καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει εκεί να επιτρέψουν πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εκεί να ε, ενταχθούν περισσότερο στην κοινότητα αξιών της Ασίας και του Ειρηνικού. Θα πρέπει λοιπόν οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν ώστε σύντομα να έχουμε την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τρόπο διαφανή. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, δύο σύγχρονε χώρε, δημοκρατικέ, από τι πιο προχμένε στον κόσμο, είναι χώρε που τι θέλουμε για εταίρου μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριο Μαριά. κύριε πρόεδρε η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου της ευρωπαϊκής ένωσης με την αυστραλία και τη νέα ζηλανδία θα οδηγήσει στην εξάλληψη των τελωνιακών δασμών με αποτέλεσμα η ένωση να πλημμυρίσει από εισαγόμενα γεωργικά κτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα σε μια φάση που οι έλληνες αγρότες οι γάλλοι και οι υπόλοιποι αγρότες της ευρωπαϊκής ένωσης κυριολεκτικά δίνουν αγώνα επιβίωσης επιπλέον η συμφωνία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα συμφέροντα των πολυεθνικών σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ένωσης τη στιγμή που οι μικρομεσαίες χυμάζονται λόγω της ίδιας της οικονομικής κρίσης και της μερκελικής λιτότητας που έχει καθυλώσει τη ζήτηση και την κατανάλωση. Ε, επίσης η συμφωνία δίνει το δικαίωμα στις πολυεθνικές να ζητήσουν αποζημίωση από τις χώρες μέλη της ένωσης στις οποίες δραστηριοποιούνται σε περίπτωση δίθεν παραβίασης των δικαιωμάτων τους επομένως θεωρώ ότι για όσο διάστημα η ευρωπαϊκή ένωση έχει τεράστιες στρατιές ανέργων το άνοιγμα των αγορών και η εμβάθυνση της παγκοσμιοποίησης μάλλον θα αυξήσει τη φτώχεια και την ανεργία στην ένωση παρά θα βοηθήσει την ανάπτυξη. ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος ε, εμπορικός εταίρος κατά σειρά της Αυστραλίας και ο τρίτος της Νέας Ζηλανδίας. Συγχρόνως η Αυστραλία είναι ο 16ος εμπορικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 51ος η Νέα Ζηλανδία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων με τις δύο αυτές χώρες. Η Συμφωνία Ελευθέρω είναι το λογικό επόμενο βήμα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι πολύ περισσότερο μάλιστα, διότι αν λάβουμε υπόψη την πίεση της Κίνας η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται <clears throat> να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις δύο αυτές αγορές. Εάν λοιπόν ξεκινήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια από ότι στην διαπραγμάτευση TTIP ώστε ότι οι πολίτες μας να ξέρουν ποιες είναι οι θετικές αλλά και οι αρνητικές επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω για την άδεξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων των Επιτροπών. Δύο σημεία όμως. Πρώτον, κάποιοι ε, τομείς ε, της γεωργικής βιομηχανίας ανησυχούν και το καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, οι ευαισθησίες τους και υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να σας πω όμως ότι όλοι έχουν να κερδίσουν. Εξίσου θα μοιραστούν τα ωφέλη δύο πλευρές. Δεύτερον, η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά πολλά περισσότερα. Δηλαδή πρόκειται για κοινέ αξίες και ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς και ιστορικούς όμως δεσμούς που θα έπρεπε να είχαν αναγνωριστεί πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό και ζητώ από την Κομισιόν να προχωρήσει τάχιστα ε, στην ολοκλήρωση αυτή τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ολοκληρώνεται η διαδικασία προσέλκυση προσοχή του Προέδρου. Κάτσε διά, κύριε Μίμητσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές. θα ήθελα να επαναλάβω την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει τα επόμενα βήματα για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. Κατά αυτόν τον τρόπο θα τηρήσουμε του κανόνες, τι πρακτικέ και θα προετοιμάσουμε τη μελέτη αντικτύπου και θα προβούμε και σε όλα τα άλλα τα προπαρασκευαστικά ε, μέτρα, ε, κάποιες διαδικασίες ε, διερεύνησης κτλ ακολουθώντας το αίτημα του Συμβουλίου για επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων. Έχουμε αναφέρει τη νέα μας πολιτική στην ανακοίνωση Trade for All, η οποία δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο Οκτώβρη. Η ανακοίνωση αυτή αναφέρει τις δεσμεύσεις μας ε, και την προσέγγιση που προτείνουμε για σημαντικά ζητήματα όπως το εμπόριο και η βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τα θέματα που αφορούν την εργασία και το περιβάλλον, τις δημόσιες υπηρεσίες και για την επίλυση ε, διαφορών ε, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Με λόγο να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, έχουμε ένα σαφή οδικό χάρτη για αυτές τις συμφωνίες και αυτό αυτόν τον χάρτη θα επιδιώξουμε να πετύχουμε με τις διαπραγματεύσεις αυτές, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία διαπραγμάτευσης είμαστε δεσμευμένοι ε, στην ε, εξασφάλιση της διαφάνειας των διαπραγματεύσεων ε, και στην πληροφόρηση, στην ανάλυση και το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά θα καθοδηγήσουν, θα είναι ο γνώμονας της δουλειάς μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.